Καλημέρα συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε μια κοινή λίμπε φάμ σε άλλη αίθουσα για την ε, ε σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που καθυστέρησε. Συγγνώμη λοιπόν για την καθυστέρηση. Συγγνώμη λοιπόν. Να ξεκινήσουμε με την έκθεση μερικής διάταξης. Υπάρχουν οι εξή αλλαγέ στο σχέδιο τη μερική διάταξη. Το 24 η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βίτσα, τον Έλληνα Υπουργό πρέπει να αναβληθεί. Θα βάλουμε ένα νέο σημείο 24, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης για την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένιον για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Θα γίνει λοιπόν αύριο 9.30 με 10 ένα νέο σημείο 24 για το θέμα της γραπτής απάντησης για τον ε, Ιταλικό νόμο για τις ε, περιόδους ε, κράτησης για τις τηλεπικοινωνίες θα γίνει αύριο στις 10 και η κοινή ψηφοφορία Λίμπε για τις εκθέσεις Μίναρ και Χάμιλτον. Α, συγγνώμη, αυτό, αυτά έγιναν. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, όπως τροποποιήθηκε, εγκρίθηκε. Λοιπόν, τι γλώσσες έχουμε. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από τα Ιρλανδικά. Λοιπόν, έγκριση των συστάσεων των ε, συντονιστών ε, εισηγητές. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ θα είναι ο εισηγητής μας για το κοινωνικό, κοινοτικό κώδικα για τις ε, βίζες. Εγώ ως πρόεδρος και λόγω μιας ανακοίνωσης της ΚΟΕ γιατί δεν είναι σε θέση να ορίσουν εισηγητή για το θέμα αυτό, θα αναλάβω την έκθεση για την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη Συμφωνία Ένωσης και Ελβετικής Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας για τους συμπληρωματικούς κανόνες για τη χρηματοδότηση των εξωτερικών συνόρων και των προξενικών θεωρήσεων. Συμφωνεί η Επιτροπή μας με αυτές τις συστάσεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Οπότε, συγγνώμη, είναι πολλές ανακοινώσεις. Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σας τα διαβάσω όλα αυτά. Κοιτάξτε τα email σας όσο το κάνω. Όχι, όχι, να μην το κάνετε, όχι, να ακούτε τι σας λέω. Λοιπόν, έχουμε δύο διορθώσεις με, βάση τον, το άρθρο 231. Πρώτη διορθώση στον κανονισμό 679 του 16 Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27 Απριλίου για την προστασία των ατόμων όσον αφορά τη διαδικασία επεξεργασίας ε, προσωπικών στοιχείων και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών στοιχείων και την κατάργηση του 3546 Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο Γενικό Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων και για την Οδηγία 216-1680 Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και πάλι 27 Απριλίου του 2016 για την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα διορθωτικά, συνάδελφοι, διορθώνουν ε, αρκετά προφανή λάθη και για να υπάρχει ε, ε, ορολογική συνέπεια. Τα έχουν κάνει οι, οι ειδικοί νομομαθείς μεταφραστές του Συμβουλίου. Έχουν καθοριστεί κάποια λάθη και γι' αυτό θα κάνουμε τις αναγκαίες διορθώσεις και θα τις αποστείλουμε στις αναγκαίες επιτροπές. Εκτός αν μία ε, πολιτική ομάδα ή ε, ορισμένοι συνάδελφοι που να είναι αρκετοί για να φτάσουν στο κατόφλι με βάση τον κανόνα 102-31 θα θεωρηθεί ότι ενεκρίθησαν αυτές οι διορθώσεις. Θέλει κανείς οι διορθώσεις αυτές να μπουν σε ψηφοφορία. Όχι. Ωραία. Οπότε εγκρίνονται αυτά τα διορθωτικά. Το επόμενο είναι η κατεξιοδότηση και πράξεις και οι εφαρμοστικές πράξεις. Λάβαμε μία απόφαση για ε, τα στοιχεία από το σύστημα εισόδου-εξόδου. Ο βασικός είναι ο κανονισμός του 2017-226 που δημιουργεί το σύστημα εισόδου-εξόδου. Η εφαρμοστική αυτή πράξη θα ανακοινωθεί μέσω του εσωτερικού μας ενημερωτικού φυλαδίου τη 27η και αρχή Μαου θα υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν αντιρρήσει. Αν έχετε την πρόθεση να υποβάλλετε αντιρρήσει, παρακαλώ να αποστείλετε ε, πριν από τι 7 Μαου λοιπόν, τι αντιρρήσει τη. Λοιπόν, επίση, ε, θα ε, ήθελα να αποτίσω φόρο στον αποδημήσαντα κύριο Στέφανο Τζαπάλα, ο οποίο απεδίμησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας από το 1990 μέχρι το 2009. Και σας παρακαλώ ε, να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμη του κυρίου Τζαπάλα. Uh, Τέλος, συνάδελφοι. Έχουμε σήμερα μια ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 11 και αύριο στις 12. Παρακαλώ λοιπόν έχετε τις κάρτες σας μαζί σας. Ωραία. Τέλος ανακοινώσεων. Σημείο 4. Ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Παρασκευή Μίχου που δεν είναι καινούρια αλλά ακόμη σχετικά καινούρια προσφάτως ε, διοριστήσα Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Home. Ναι, είναι πρώτη φορά, ε. πρώτη φορά που είστε εδώ ως Τι συνέβη? Ε, με συγχωρείτε, ε, νομίζω ότι δεν μιλάω και δεν δυνατά. Α, δεν φταίω εγώ. Εντάξει. Okay. Όταν η κυρία Βεζιά βάζει τι φωνές ε, με τρομάζει, με ξυπνήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ωραία, τώρα έχω αρκετή αδρεναλίνη. Λοιπόν, καλωσορίζουμε την κυρία Μίχου. Βεβαίω η δουλειά της ε, είναι ιδιαίτερα απαιτητική και τη ευχόμαστε καλή τύχη κατά την υπόλοιπη θητεία μας και στο μέλλον. Για σήμερα υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα, ως συνήθως στην Επιτροπή μας αλλά για να διαμορφώσω κάπως τη συζήτηση ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για την διαλειτουργικότητα της επικείμενης προτάσεις, το πακέτο για το άσυλο και την κατάσταση στο Συμβούλιο. Όλα αυτά θα μπορούσαν να μας απασχολήσουν για ένα ολόκληρο πρωινό. Τι γίνεται με το Δουβλίνο, τον κανονισμό του Δουβλίνου. Ξέρουμε ότι έχει μπλοκαριστεί η μπλε κάρτα, η διαχείριση των συνόρων με το IPM, τα επόμενα προγράμματα. Προφανώς πολύ σημαντικά θέματα, αλλά ίσως και άλλα που θα ήθελα να θίξουν οι διάφοροι συνάδελφοι. Με χαρά λοιπόν να σας δώσω τον λόγο και πάλι σας συγχαίρω για τον διορισμό σας. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι και πάλι εδώ, στο Κοινοβούλιο. Έχω συνεργαστεί με πολλούς από εσά στο, στο παρελθόν, όταν ήμουν ακόμη στην Γενική Διεύθυνση για θέματα δικαιοσύνη. Έχω ήδη ένα μήνα στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Και έχω έρθει για να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, να ακούσω τις απόψεις σας. Έχουμε μια πολύ επικοδομητική και καλή συνεργασία με τους συγητές και την Επιτροπή σας γενικότερα και ο ρόλος μου είναι πιστεύω να συμβάλλω σε αυτή την καλή ατμόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα συνεργασίας και αυτό θα το πράξω στο μέγιστο των δυναμεών μου. Οι προτεραιότητες της Γενικής Διεύθυνσης ως προς το νομοθετικό κομμάτι είναι υψηλές η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο στη κοινή διακήρυξη των προτεραιοτήτων έχουν ορίσει ποιες είναι οι προτεραιότητες τους. Εγώ θα τοποθετηθώ σε ορισμένες από αυτές, τις προτεραιότητες της κοινή διακήρυξης. Ταυτόχρονα όμως θέλω να επισημάνω ότι πιέζει ο χρόνος, γιατί μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα μετράει, όχι κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα μετράει προκειμένου να προχωρήσουν οι τελικές συμφωνίες να είμαστε έτοιμοι μέχρι το Μάιο του 19. Οι κύριες προκλήσεις λοιπόν που έχουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου. Πρόκειται για θέμα προτεραιότητας για μας και νομίζω προτεραιότητα υψηλή έχει μόνο για την Επιτροπή αλλά και για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Εργαζόμαστε εντατικά με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εξεύρουμε συμφωνία στα διάφορα συστατικά της ε, τελικής συμφωνίας για το κείμενο αναζητώντας τη λεπτή αυτή ισορροπία μεταξύ ευθυνών και αλληλεγγύης. Το χρονοδιάγραμμα, το φύλλο που ακολουθούμε με τους συναδέλφους. Είναι ήδη γνωστό, είναι ήδη καταγεγραμμένο στο θεματολόγιο των ηγετών, δηλαδή εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέλουμε να έχουμε μια γενική πολιτική προσέγγιση και καθοδήγηση για το τι θα κάνουμε περαιτέρω. Και δέσμευση πως η δουλειά μας ακολουθεί την ορθή κατεύθυνση. Η Βουλγαρική Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει μορφή σε αυτές τις προτάσεις. Ε, οι συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετικές, πάντως υπάρχει πλήρης υποστήριξη από πλευράς της Επιτροπής στις προσπάθειες της Προεδρίας, της Βουλγαρικής Προεδρίας, μέχρι τις 15 Μαΐου που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να καταθέσουμε το φάκελο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διανύουμε μία κρίσιμη περίοδο, κρίσιμη γιατί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με το κείμενο, με όλο το φάκελο, όπως θα κατατεθεί τελικά στο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 Μαΐου. Πριν από δύο-τρεις εβδομάδες που συνάντησα τον πρόεδρο, τον διαβεβαίωσα ότι θα παραμείνω στη διάθεση του Κοινοβουλίου και θα έρθω και στην Επιτροπή για να συζητήσουμε το πλήρες πακέτο προτάσεων, την πλήρη με προτάσεων για το άσυλο, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό βέβαια το τμήμα της ε, διαδικασίας αυτής του θέμα του Δουβλίνου, αλλά είναι ένα σύνολο οι δέσμοι προτάσεων για το άσυλο και πρέπει μαζί να το κλείσουμε. Να την κλείσουμε. Eurodac. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα στο Κοινοβούλιο, αλλά είναι και μεγάλη μέρα στο Κοινοβούλιο, γιατί θα είμαι το απόγευμα σε αντίστοιχη συνεδρίαση. Ε, είμαστε πολύ κοντά λοιπόν σε συμβιβασμό και έχουμε σήμερα τριμερή διάλογο. Ο εισηγητής με τους κοιόδης εισηγητές έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχουν τη συνεδρία προπαρασκευής για την απογευματινή τριμερή. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η αναθεωρημένη Eurodac ξεπερνά το πεδίο της μεταρρύθμισης ε, του θέματος του ασύλου. Και γι' αυτό και η ανακοίνωση και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τονίζουν ότι η Eurodac και ο αναθεωρημένος κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια ενιαία δέσμη. μπορούν να προχωρήσει το κάθε θέμα χωριστά σε σχέση με το υπόλοιπο πακέτο του ασύλου. Η Eurodac λοιπόν έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα των επαναπατρισμών αλλά και την αναγνώριση ανηλίκων που δεν έχουν καταγραφεί σε καμία βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα θα βοηθήσει στη διαλειτουργικότητα και συνεργασία με άλλα συστήματα δεδομένων όπου αυτό είναι απαραίτητο. Άλλη πρόταση που έχει προχωρήσει ικανοποιητικά μέσα από τις συζητήσει, είναι ο κανονισμός για την υποδοχή και την εγκατάσταση κανονισμός πλαίσιο. Ε, οι τριμερείς συναντήσεις πήγαν πολύ καλά, είμαι πολύ ικανοποιημένη από την πρόοδο. Η κυρία Φαγιώκη, και η Νετφέλτ ε, και η κυρία Μποκ έχουν βοηθήσει σημαντικά ως εισηγήτρια και συνεισηγήτριες στην εξέβρεση συμβιβαστική λύσεως ε, και σε επίπεδο Συμβουλίου υπό την Βουλγαρική Προεδρία. Ωστόσο, θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερε προσπάθειες και εδώ έχουμε να κάνουμε τον κανονισμό διαδικασιών για το άσυλο, όπου δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί εντολή για διαπραγμάτευση. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Κορεπέρ τόνισα στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται εντατικά για την εντολή αυτή. Γιατί αυτή η διαδικασία, ο κανονισμός δηλαδή για τη διαδικασία ασύλου, είναι κομμάτι της δέσμης για το άσυλο και θα έχει κρίσιμη σημασία όταν θα έρθει η ώρα να ε, υλοποιηθεί το Δουβλίνο, όταν θα έρθει η ώρα να αξιοποιήσουμε ε, αποτελεσματικές διαδικασίες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτόν τον κανονισμό και θα απευθυνθώ στην κυρία Φερέρα και τους, ε, την εισηγήτρια και τους συνεισηγητές για να προσφέρω τις υπηρεσίες και την ε, ε, αρρωγή μου εάν και εφόσον αυτό χρειάζεται. Στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης ανέφερε κάποιες ε, νέες προτάσεις ο Πρόεδρος. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Προσπαθούμε πάντως και τώρα ακόμα να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις διαπραγμάτευσης για συμφωνία με τα κράτη-μέλη, στο βαθμό που μπορούμε, να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, γιατί ξέρω ότι ήταν και δική σας προτεραιότητα το θέμα αυτό της Επιτροπής σας δηλαδή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης, ορίζουμε πιλωτικά προγράμματα για την νόμιμη μετανάστευση, νομότυπη μετανάστευση και κυρίως από την Αφρική ε, μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με, με νομότυπη εξέβρεση εργασίας κτλ. Οικονομική στήριξη θα προσφέρουμε, τα, τα πιλωτικά αυτά προγράμματα μπορεί να βρίσκονται τώρα σε μια πρώιμη φάση αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία δηλαδή. Τώρα θα περάσω στην ε, προξενική θεώρηση. Είστε ενήμεροι για την ε, πρόταση που καταθέσαμε το Μάρτιο, που στόχο έχει να ενισχύσει την πολιτική της προξενικής θεώρησης, να την καταστήσει πιο ασφαλή και πιο αποτελεσματική. Ε, χρειάζεται, και αυτός είναι και ένας από τους στόχους της πρότασης, να υπάρξει μια κοινή πολιτική προξενικών θεωρήσεων που θα στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση του επαναπατρισμού παράτυπων μεταναστών. Μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα συμπληρωθεί η πρόταση αυτή με το σύστημα πληροφοριών προξενική θεώρησης που θα έρθει το Μάιο και βεβαίως θα είμαστε στη θέση σας για να το συζητήσουμε. Διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα ήταν ε, και παραμένει ε, θέμα προτεραιότητας, παραμένει θέμα προτεραιότητας και για τις διαπραγματεύσει. Η Βουλγαρική Προεδρία στοχεύει σε μια γενική προσέγγιση. Αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλη είναι η κλίμακα του έργου που έχουμε αναλάβει. Είμαι βεβαία όμως ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να, η θα είναι σε θέση να υιοθετήσει θέσεις πριν από το... η Επιτροπή μας θα είναι σε θέση να υιοθετήσει θέσεις πριν από το καλοκαίρι ώστε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Αυστριακή Προεδρία. Σας είπα ε, τα θέματα αυτά ποια είναι και οι προτεραιότητες, αλλά για μένα προσωπικά θέλω να επισημάνω όταν ήμουν ακόμη αναπληρώτρια γενική διευθύντρια ότι ήταν στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου και γι' αυτό με ενδιαφέρει προσωπικό, στο EDPS και το και η Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα έχουν εμπλακεί εξ αρχής σε κάθε φάση της προετοιμασίας για τις προτάσεις αυτές, όπως επίσης και ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου, Όπως είπα, η DPS και η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ήταν ε, μαζί με αυτούς στις συνομιλίες, στην προετοιμασία. Είμαι ευγνώμων για τη δουλειά που βλέπω ότι προχωρεί και τις θέσεις τους που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, θέσεις οι οποίες και θα ε, αξιοποιηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις. Έχουν οριστεί από ό,τι γνωρίζω εδώ οι συγητές σας, ο κύριος Λέναρς, ο κύριος Μελό και οι λοιποί συνεισηγητές και με χαρά θα συνεργαστώ μαζί τους. Το ΕΝΤΕΑΕΣ έχει προχωρήσει πολύ καλά πιστεύω από ό,τι μαθαίνω. Έγινε σήμερα το πρωί συζήτηση για μια συμφωνία ε, για αναθεωρημένη ως προσωρισμένα μόνο μια εντολή και είμαι βεβαία πως το συμβαστικό κείμενο που θα κατατεθεί στη συνέχεια θα αντιστοιχεί και στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν 2. Νέες εξελίξεις, σημαντικές εξελίξεις, νέο κείμενο και πιστεύω ότι θα έχουμε προς τα τέλη Μαΐου το τελευταίο τριμερή διάλογο. Παρακολουθούμε συνέχεια και στηρίζουμε τις εξελίξεις στην πρόταση αυτή, όπως και στην EU ε, όπου γνωρίζω ότι υπάρχουν δύο σημεία, ή μάλλον υπήρχαν επιτάπητος δύο σημεία ακόμα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ήδη υπάρχουν εξελίξεις, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον. Ε, η μία εξέλιξη αφορά επέκταση ή και νέες εγκαταστάσεις και η δεύτερη εξέλιξη έχει να κάνει με την ε, διευκόλυνση κρατών που δεν έχουν η ικανότητα για ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών όπως εμείς τα ζητούμε, τα απαιτούμε. Ε, και σε αυτό η Λίζα, το σύστημα Λίζα θα βοηθήσει τα κράτη αυτά μέλη ώστε να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις του συστήματος. Η κυρία Μάκοβε, η συγγήτρια, πιστεύω ότι κάνει καταπληκτική δουλειά και σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν, κάπου στα μέσα Ιουνίου η Επιτροπή και ο Πρόεδρός σας ε, θα λάβει τη σχετική επιστολή. Η Επιτροπή μας λοιπόν θα καταθέσει επιστολή με τις ε, προτάσεις της που θα τροποποιούν τις προτάσεις διαλειτουργικότητας και γι' αυτό θα ήθελα να σας ε, περιγράψω λεπτομερώς το πώς θα διαμορφωθούν οι αλλαγές σε σχέση με τις διάφορες προτάσεις. Και επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι συνοριακή έλεγχη, και ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα που σας απασχολεί ιδιαίτερα, εσωτερική έλεγχη, έλεγχη στα εσωτερικά σύνορα. Αλλά ταυτόχρονα βέβαια μας, μας απασχολεί πολύ και το θέμα των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και για ορισμένα κράτη-μέλη ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα είναι προϋπόθεση για κάποια συμφωνία ή για οποιαδήποτε συμφωνία στο συνολικό πακέτο προτάσεων για το άσυλο. Για τους εσωτερικούς λοιπόν ελέγχους, ε, χτες έκανα συνάντηση με τους πρέσβεις των κρατών εκείνων που έχουν κοινοποιήσει το εξάμεινο ή και παράταση του για εσωτερικούς ελέγχους και, τα όμορα, και των ομόρων κρατών τους σε μια πολύ επικοδομητική και ειλικρινή συζήτηση για τις συνέπειες αυτών των ελέγχων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τους εξαλείψουμε. Πρέπει επίσης να σημειώσω όμως ότι είναι σημαντικός ο αντίκτυπος οικονομικός, μένα, αλλά όχι μόνο. Είναι αντίκτυπος και προς την αξιοπιστία του Σέγγεν και σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διτεθειμένη να διδραματίσει το ρόλο της έτσι ώστε να ε, αποσοβηθεί αυτός ο κίνδυνος. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος κατέστησε επίσης σαφές ότι οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα δεν μπορούν να συνεχιστούν επαόριστα. Δεν θέλω να επεκταθώ διεξοδικά στη στις προτάσεις για την ασφάλεια που υιοθετήσαμε τον Απρίλιο. Είναι πολλές όμως οι προτάσεις ε, εκτεταμένες. Έχουν ξεκινήσει συζητήσει και με την κοινωνία των πολιτών, επιχειρήσεις, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με την διευκόλυνση πρόσβασης σε οικονομικά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών. Θυμάμαι ακόμα συζητήσει που είχαμε πραγματοποιήσει σε σχέση με την, με την ευκαιρία μάλλον της οδηγίας για την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. και τη δυνατότητα παρακολούθηση των χρηματοπιστωτικών ροών. Νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ διεξοδική αξιολόγηση, όπως άλλωστε έχει γίνει και αντίστοιχη αξιολόγηση για τα λοιπά σχετικά θέματα. Επίσης έχουμε κάνει ε, πρόταση για τις ε, πρόδρομες ουσίες ή υλικά για εκρηκτικά και για τις διαδικασίες για τα πυροβόλα όπλα και συνεργασία μεταξύ των αρχών για το εμπόριο ε, πυροβόλων όπλων. Κλείνοντας όμως θα ήθελα να σταθώ λίγο στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Στις 2 Μάη με την προσεχή εβδομάδα πρόκειται να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για το Πουδουπού. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα η συζήτηση προσανατολισμών στην Επιτροπή στη συλλογική της ε, μορφή. Έχει ε, αναγνωριστεί από όλους η σημασία της διατήρησης χρηματοδότησης του τομείς αρμοδιοτήτων μας από όλους Εγώ νομίζω ότι θα διατηρηθούν τα ποσά που αφορούν το κομμάτι αυτό και μάλιστα μπορεί και να ενισχυθεί ο προπολογισμό στους τομείς που μας ενδιαφέρουν για το άσυλο αλλά και για την μετανάστευση και, τον εξωτερικό, και τα εξωτερικά μέσα γιατί όπως ξέρετε τα εξωτερικά νομοθετήματα γιατί όπως ξέρετε ε, έχουμε και ζητήματα διαχείρισης των εξωτερικών μεταναστευτικών ροών που καλύπτονται από αυτά. Μέσα στις δυσκολίες τις μεγάλες που αντιμετωπίσαμε στην κρίση μετά το 2015, κατέστησα θέση ότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνο μία εσωτερική προσέγγιση. Δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Πρέπει βεβαίως και να επιδειχθεί ε, υπευθυνότητα. Πρέπει να επιδειχθεί και αλληλεγγύη, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να τίνουμε και χείρα βοηθεία προ τι χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντα να εξεύρουμε τι κατάλληλε λύσει, προσφέροντα άσυλο μεν και προστασία σε όλου αυτού που το έχουν ανάγκη. Ταυτόχρονα όμω και μεριμνώντα έτσι ώστε εκείνοι οι οποίοι δεν χρήζουν προστασία ε, και βρίσκονται στην Ευρώπη να μπορούν να επαναπατριστούν με ασφάλεια στις χώρες τους και σε αυτό θα δώσουμε σημαντικά χρηματικά ποσά. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Στηρίζομαι σε εσά, στηρίζομαι στη συνεργασία. με την Επιτροπή σας. Εάν κάτι δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω σήμερα, πολύ ευχαρίστω. Σας διαβεβαιώνω, θα επανέλθω και γραπτός. Ευχαριστώ. Μάλλον θα πρέπει να γίνει αυτό γιατί πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ένα θέμα το οποίο θα το θέσω άμεσα αναφερθεί. Υπάρχουν ε, ε, δύο, δύο σκιώδεις οι οποίοι θα πάρουν το λόγο. Για την μπλε κάρτα, ναι. σχετικά με την μπλε κάρτα παραμονής. Είναι αλήθεια ότι και ε, τα πράγματα εξελίσσονται γρήγορα. Δεν έχει υπάρξει, δεν έχει προχωρήσει η εναρμόνιση του συστήματος. Ο λαϊκισμός και οι εσωτερικές ε, νομικές ρυθμίσεις ε, υπό την πίεση του λαϊκισμού και σε χώρες όπως η Γερμανία δεν έχουν βοηθήσει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε σε σχέση με τις προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Αν μπορέσουμε λοιπόν να βρούμε κάποιον τρόπο να προχωρήσουμε, έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λειτουργήσει προοδευτικά, ασκεί κριτική σε νέους κανόνες όταν είναι αντίθετη με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αρκετά με την προφανή πλέον υποκρισία Λοιπόν, η κυρία Σίπολ, παρακαλώ μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συγκεντρωθώ σε συγκεκριμένα θέματα για τη διαλειτουργικότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να βιαστούμε. Η βασική ιδέα είναι ότι δεν κάνουμε κάτι το δύσκολο, απλά προσπαθούμε να συνδέσουμε τις διαθέσιμες νομικές βάσεις έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ε, σε πολύ περισσότερες από μία βάση δεδομένων και να εκδίδεται το έγγραφο πολύ πιο γρήγορα. Αλλά δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την πρόσταση και την προσ... με πρόσβαση και την προστασία των δεδομένων. Γιατί να βιαστούμε να τελειώσουμε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και μετά να συζητήσουμε τις πρακτικές επιπτώσεις. Δεν μου αρέσει αυτό. Για το πακέτο για το άσυλο είπατε ότι το Eurodac δεν θα πρέπει να συναποτελέσει τμήμα του πακέτου. Ενώ πραγματικά θα ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι στο τέλος θα έχουμε το Eurodac, αλλά τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν, σαν παράδειγμα, να βρούνε κάποια λύση για το Δουβλίνο. Συνεπώς λοιπόν είναι πολιτική απόφαση αν θα κάνουμε πακέτο ή αν θα το αφήσουμε εκτός. Ε, αλλιώς το Δουβλίνο ας πούμε δεν θα τεθεί ποτέ προς συζήτηση και δεν θα βρει λύση. Τώρα για τα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα. Πήρα το μήνυμα από τον Επίτροπο Αβραμόπουλο ότι οι έλεγχοι στα εξωτερικά θα πρέπει να διονίζονται. Ή μάλλον τα, ε, στα εσωτερικά σύνορα. Μα ε, δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο και όμως όμως συμβαίνουν σε ορισμένες περιπτώσεις. Ε, διαρωτώ με πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία Ποια είναι η βασική ιδέα, όλα τα σύνορα θα είναι κλειστά. Λοιπόν, ε, λέμε ότι δεν θα πρέπει να κρατήσει η κατάσταση αυτή περισσότερο, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά υποχωρεί. Τώρα για τα υπόλοιπα καταπιστεύματα τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τελικά κάποιες ε, ιδέες μετά τα αιτήματα των κρατών μελών, το τι θα πρέπει να δώσει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Έχει κάποια ιδέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες μας. Ναταλή Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Κλόντ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και τα πιο σημαντικά θέματα έχουν ήδη τεθεί από την κυρία Μίχου. Τρία σημεία σύντομα, τα οποία άπτονται των σημείων ε, ε, ρήξης, αν θέλετε. Για την μπλε κάρτα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, Είμαστε πολλοί στους σκιώδεις που πιστεύουν ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από την υποκρισία και θα πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Δεν μπορούμε στην Ευρώπη εμείς να εξηγούμε ότι θα πρέπει να είμαστε δεκτικοί σε σχέση με τις ε, ειδικέ μεταναστευτικές ροές, ε, με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες ικανότητες και θα συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ ταυτόχρονα στις συναντήσεις μας ε, να ακολουθούμε μια πρακτική πλήρους αποκλεισμού έβρεσης λύσης. Συνεπώς λοιπόν ε, θα πρέπει να βρούμε μια διαφορετική λύση, ίσως αυτή την οποία προτείνει ο Κλοντ για να προχωρήσει το θέμα έχει την στήριξη πολλών σκιωδών επί του θέματος αυτού, το οποίο δυστυχώς κρατάει πολύ. Τώρα για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, κυρία μου, αναφερθήκατε στην ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος, απ' την άλλη βλέπουμε ότι έχουν μπλοκάρει τα πράγματα, θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να ξεπεραστεί η δυσκολία, γιατί είναι μια δυσκολία η οποία επηρεάζει άμεσα τους Ευρωπαίους πολίτες. Και το τρίτο θέμα, το οποίο δεν αναφέρθηκε, αναφέρεται στο, στο πάγωμα και στην κατάσχεση των προϊόντων παράνομων εσόδων. Είναι ένας δρόμος που θα βοηθήσει στην έβρεση αποζημίωσης για τα θύματα και που θα επιτρέψει επίσης να εισπραχθούν και πολλά, πολλά χρήματα για να αποζημιωθούν όπως είπα τα θύματα. Και εδώ δεν έχει υπάρξει λύση και γι' αυτό θα ήθελα να εμείνετε έτσι ώστε να βρεθεί τελικά κάποια λύση. Judith Αργεντίνη. Εκπλήσωμαι ή μάλλον αναρωτιέμαι τι θα προσφέρει το Συμβούλιο του Ιουνίου και ιδιαίτερα η προθεσμία αυτή μέχρι τις 15 Μαΐου είναι κάτι το οποίο με μπερδεύει. Ε, να επαναλάβω αυτό που ακούστηκε, ότι σε σχέση με το άσυλο με τη μετανάστευση έχουμε να κάνουμε με πακέτο. Εγώ βγήκα έξω από την συνάντηση των σκιωδών για το Eurodac για να έρθω εδώ και το θέμα είναι αν μπορούμε να πιέσουμε να, ε, τα παιδιά να δώσουν ε, τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Αυτό δεν βοηθάει την ευημερία των παιδιών, δεν έχει σχέση με το άσυλο που μπορεί να αιτηθούν, αλλά έχει κάτι το εντελώς διαφορετικό σαν σκεπτικό. Και θα μπορούσα να καταλάβω ότι το Eurodac δεν θα είναι τμήμα του πακέτου, αλλά θα ήθελα η μπλε κάρτα και άλλες πρωτοβουλίες στο μέλλον για την νόμιμη μετανάστευση να γίνουν επιτέλους αντικείμενο συζήτηση, όπως επίσης και να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την επανεγκατάσταση και θα πρέπει η Επιτροπή να στείλει το μήνυμα στο Συμβούλιο ότι το άσυλο και η μετανάστευση αποτελούν ένα σύνολο πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώς δεν θα μπορούμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα σταματώντας και βάζοντας επιπλέον σημεία ελέγχου. Τώρα, το θέμα είναι τι κρίση έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ε, κλείνει η Δυτική Ευρώπη, τα κέντρα ετούν τον άσυλο. Ε, απομακρύνουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, και όταν αρχίζουν να χρησιμοποιούν ε, νέους δρόμους, όταν προσπαθούν να διασχίσουν τον ποταμό για να περάσουν στην Ελλάδα και όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι δεν μπορείτε να έχετε στα νησιά περίκλειστους ε, τους πρόσφυγες, θα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ε, κοιτάξτε, έτσι και αλλιώ περιμέναμε μια τέτοια απόφαση. Είναι, είναι λογική μια τέτοια απόφαση και αυτός ο ο γεωαποκλεισμός δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί επί μακρόν. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να στηρίξουμε το σύνολο του πακέτου που είναι η θέση του Κοινοβουλίου γιατί αν υπακούσουμε στις επιθυμίες ε, του ε, Συμβουλίου και της Βουλγαρικής Προεδρίας η οποία βλέπει τα θέματα του ασύλου και της μετανάστευσης με ιδιαίτερα κατασταλτικό τρόπο τότε δεν θα περάσουμε τις απόψεις μας. Κοιτάξτε παρακαλώ, ε, θέλουμε να πάρουμε μια απάντηση από την κυρία Μίχου και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τέσσερις οι ομιλητές, να είστε παρακαλώ σύντομοι. Σπινέλη, Γκραπίνη, Βεργιά και Γκόμες. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να εμβαθύνω εδώ σε αυτό το οποίο είπατε για την παράλυση των διαπραγματεύσεων για την μπλε κάρτα. Ω κοιόδηση συγγήτρια για τη μεταρρύθμιση θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου αλλά και τη δυστημία μου για την παράλυση αυτή η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην ανικανότητα του Συμβουλίου να κάνει επικοδομητικό διάλογο με το Κοινοβούλιο μια ανικανότητα η οποία μετετράπει μέσα στο χρόνο σε έλλειψη ε, βούλησης. Να θυμίσω δύο στοιχεία εδώ. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης εγώ υποστήριξα και η πολιτική μας ομάδα υποστήριξε επίσης τον εισηγητή, την εισηγήτρια, ο οποίος με πάρα πολύ διπλωματικότητα προχώρησε, διετήτευσε, προώθησε θέσεις προς το Συμβούλιο και σε ακαθόδη κυρίως θέματα. Κάποιες από τις κόκκινες γραμμές μας παραμένουν ε, με πρώτη και καλύτερη την εναρμόνιση. Εμείς θελήσαμε να υπάρξει μια πιο ελαστική και σταδιακή εφαρμογή. Επίσης ε, δείξαμε την, την ευελιξία από πλευράς μας από την άλλη όμως το Συμβούλιο δεν γίνεται τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Το Συμβούλιο στην ουσία είπε ότι θέλει να διαπραγματευτεί μια οδηγία χωρίς ουδεμία προστιθέμενη αξία σε σχέση με την ισχύουσα. Αρνείται την εναρμόνιση. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο πρόεδρος Μωράης, να μην συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, ε, γιατί έτσι θα καταλήξουμε σε ένα εντελώς νέο κείμενο, εντελώς στρεβλό. Και τώρα, δυστυχώς, η πολιτική του ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια καταστροφική πορεία. Το ότι δεν μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία, ακόμα και κατελάχιστον, κατελάχιστον σε σχέση με τους νόμιμους τρόπους μετανάστευσης είναι πραγματικά σύμπτωμα βαριάς ασθένειας στην ευρωπαϊκή πολιτική που θα υπονομεύσει το δημογραφικό μέλλον της Υπήρου μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα στην κυρία Διευθύντρια. Κάποια από τα στοιχεία τα οποία εμείς πρεσβεύουμε συμφωνούν με αυτά τα οποία λέτε εσείς κάποια. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να πιέσουμε επιτέλους το Συμβούλιο και να το βγάλουμε από αυτό το αδιέξοδο. Τι επιχειρήματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να σταθείτε πιο αποτελεσματικοί από ό,τι εμάς και από ό,τι ο Κλοντ κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ Μπάμπρα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις, γι' αυτό παρακαλώ να είστε όσο ο πιο σύντομοι μπορείτε. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Πολλά έχουν υποθεί και συμφωνώ απόλυτα με όσα υπόθηκαν. Μια σύντομη λοιπόν ερώτηση. Σας ευχαριστώ για αυτό που μας είπατε. Και θα ασχοληθώ λοιπόν με τα εξής. Είπατε ότι μέχρι τις 15 Μαΐου θέλετε να έχετε κρίνει ένα κείμενο που θα υποβάλλετε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και εν ώψη των ε, μελλοντικών εκλογών πρέπει να καταλάβετε ότι η κοινή γνώμη αλλά και οι αρχές στα κράτη-μέλη δεν κατανοούν ε, τη σημασία του θέματος της μετανάστευσης και της αντιμετώπισης του. Πρέπει να έχουμε ένα σαφές μήνυμα να αποστείλουμε στους πολίτες. Πρέπει το Συμβούλιο να υιοθετήσει σαφή άποψη. Τι μπορείτε να κάνετε περισσότερο για τον κανονισμό, για τη διαδικασία του ασύλου. Και θέλουμε να δούμε το κείμενο που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο στις 15 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος, η κυρία Βεωζία. Θα επιχειρήσω να είμαι ταχύτατη. Α, γιατί θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να το συζητήσουμε, γιατί θίξατε πολλά θέματα. Και σας ευχαριστώ. Είπατε ότι πολλά από αυτά τα θέματα ήταν προτεραιότητες για τα τρία θεσμικά όργανα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είμαι πεπισμένη ότι τελικά ε, τα τρία θεσμικά όργανα έχουν τις ίδιες προτεραιότητες τελικά. Όλα αυτά είναι προτεραιότητες. Γι' αυτό έχουν υπάρξει ε, αδιέξοδα σε διάφορα θέματα και το θέμα δεν είναι να έχουμε συμφωνία πάση θυσία για κάποια, αν αυτό σημαίνει υποχώρηση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν είπατε πολλά, κυρία μου, για το θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου. Καλύτερα να πω ότι δεν άκουσα τίποτα για αυτά, που είναι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ιδιαίτερα πολλά θέματα τα οποία αναφέρατε. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ ε, υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Καλά. Αλλά πρέπει επίση να υπάρχει και η αρχή τη αναλογικότητα και αναγκαιότητα μεταξύ τη ε, ανάγκη για ασφάλεια και του σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην ομιλία σα, όπω και αυτά που ακούω από τα κράτη-μέλη, και συγγνώμη που σα το λέω, υπάρχει μια αιμονή ιδέα για αυτό που λέτε η παράνομη μετανάστευση. Για μας και για πολλού άλλου εδώ δεν υπάρχει παράνομο μετανάστε. Δεν υπάρχει κανένα παράνομο μετανάστε. Υπάρχουν μετανάστε που είναι σε παράτυπη κατάσταση γιατί η νομοθεσία της Ένωσης και των κρατών μελών τους βάζουν σε αυτή την παράτυπη θέση. Θα έπρεπε λοιπόν να ξαναθέσουμε το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του σεβασμού του δικαιώματος, του δικαιώματος ασύλου, της ε, της Γενέβης, να είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Γαλλία υπάρχει ένας Ιρανός αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι σε κέντρο κράτησης, ο οποίος απειλείται με απέλαση ανα πάσα στιγμή, ενώ είναι καταδικασμένος σε θάνατο στη χώρα του. Καταδικασμένος σε θάνατο. Ε, Βεβαίω έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα στη Γαλλία, αλλά είναι καταδικασμένο σε θάνατο στο Ιράν γιατί είναι χριστιανό. Τι παριστάνουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πρόκειται να στείλουμε πίσω στο Ιράν κάποιον ο οποίο είναι καταδικαμένο σε θάνατο λόγω της θρησκείας του. Νομίζω ότι φτάνουμε πραγματικά στα όρια, στα όρια του απαράδεκτου. Και θα πρέπει να παρακολουθούμε και να μελετάμε τέτοιες καταστάσεις πολύ ε, προσεκτικά. Και η τελευταία, η κυρία Ανακόμες παρακαλώ σύντομα, κυρία Μίχου, λέει η κυρία Γκόμες. Με συγχωρείτε, καθυστέρησα, δεν μπόρεσα να σας ακούσω. Αλλά ελπίζω ότι θα σας ακούσω σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω. Πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση όχι μόνο με εμά, αλλά και στην ε, σχέση της με τα κράτη-μέλη. Ε, δεν είναι ο ρόλος σας να τους λέτε την αλήθεια. Επειδή ακριβώς δεν επιτρέπουν ε, ασφαλή είσοδο σε πρόσφυγες και μετανάστες, επειδή δεν συμφωνούν για το Δουβλίνο για να προχωρήσει η μπλε κάρτα, στην ουσία εμείς, εμείς δίνουμε δουλειά στους διακινητές. Αυτό είναι η αλήθεια, αυτό πρέπει να πείτε στα κράτη-μέλη και όχι να συμφωνείτε με την ρητορία τους περί ε, ε, στην, στο Σουδάν και στην Τουρκία. Και η υποκρισία είναι στον κολοφόνα της. Όταν τα κράτη-μέλη πουλάνε πρόσβαση στον χώρο Σέγγεν, σε ορισμένους, ή ακόμη και διαβατήρια. Υπάρχει μια έκθεση το Νοέμβριο. Ε, περιμένουμε να την ε, ε, δώσει, να μας τη στείλει η Επίτροπος Γιούροβα τον Νοέμβριο, αυτές τις ιστορίες για τις χρυσές βίζες. Αλλά φυσικά ε, δεν έχει καμία έννοια. Είναι τρομερές οι αντιφάσεις. Θα πρέπει να γυρίσουμε στο θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, με μια συγγνώμη ταυτόχρονα προς την κυρία Μίχου, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε σε όλα τα ζητήματα. Πέντε λεπτάκια, Τάνια, συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, αλλά έχουμε μακρές ψηφοφορίε, αρχίζουν να γίνανε συνάδελφοι. Πάντα βέβαια ε, και όλα αυτά με την επιφύλαξη ότι ε, θα σας ξαναδούμε και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Δώστε μας λοιπόν κάποιες ε, λακωνικές απαντήσεις και όπως είπαμε και έγραπτος, αλλά και σε μια επόμενη ευκαιρία συνεδρίασης θα τα ξαναπούμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικά τα θέματα και εν εξελίξει μάλιστα. Δώστε μας όμως κάποιες επιγραμματικές απαντήσεις. Η κυρία Μίχου, πολύ ευχαρίστω να συζητήσω μαζί σας όλα τα θέματα που αναφέρατε και εσείς όπως και εγώ ε, Πώ είπαμε, δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειε σήμερα, αλλά θα τα πούμε. Αυτή η άδεια παραμονής, η μπλε κάρτα, το έχουμε συζητήσει μαζί σας και γι' αυτό και καταθέσαμε τις προτάσεις. Προσπαθήσαμε να ε, επιτελέσουμε το ρόλο μας ως θεσμικού οργάνου, κάνοντας προτάσεις που δεν θα ήταν ε, γράμμα κενό και γι' αυτό έχει παγώσει προς το παρόν αυτή η υπόθεση. Δεν λέω ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να βρούμε ευκαιρίες και πρέπει εγώ να βρω την ευκαιρία. Γιατί δεν είχα το χρόνο από την ανάληψη της Γενικής Διεύθυνσης ε, Home να αναζητήσω λύσεις. Γιατί εάν δεν βρεθούν λύσεις, γράμμα κενό δεν είμαι διατεθειμένη να καταθέσω. Τόσο απλά τα πράγματα. Για το άσυλο. Συμφωνεί η Επιτροπή μας, όπω και εγώ προσωπικώ, ότι πρέπει να έχουμε μια ε, γενική και ολιστική προσέγγιση στη δέσμη των ε, μέτρων για το άσυλο, αλλά δεν ε, έβγαλε από το πακέτο τη Eurodac η Βουλγαρική Προεδρία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποφάσισε ότι είναι δυνατόν να ε, εξεταστεί και να προχωρήσει χωριστά το θέμα της Eurodac λόγω και της λειτουργικότητας που προσφέρει σε διάφορες άλλες λύσεις. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω και θα γίνει πολύ το σεβαστό αυτό το οποίο θα αποφασίσετε. Αλλά αυτό δεν θα μας εμποδίσει εμάς να αναζητήσουμε συμβασμούς και λύσεις που θα φέρουν αποτελέσματα και θα χτίσουν κομμάτι-κομμάτι τις διάφορες δέσμες. Δεν μπορώ να συμφωνήσω δηλαδή με τα κράτη-μέλη ή με εκείνους που λένε ότι α, το Δουβλίνο δεν το θέλω, την αλληλεγγύη δεν τη θέλω, Θέλω ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα. Όχι, δεν μπορεί να πάει έτσι. Πρέπει να είναι ολιστική η προσέγγιση. Όμως η Eurodac για μας, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναλαμβάνω, δεν είναι στοιχείο εκ των ουκάνευ για τη δέσμη. Αλλά θα το αποφασίσετε εσείς. Διαλειτουργικότητα. Είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμη σημασία θέμα. Μπορούμε να συστήσουμε τις λεπτομέρειές της, όχι τώρα βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντική δέσμη και κρίσιμη, διότι θα δώσει την ε, διασύνδεση όχι μόνο πολιτική αλλά και πρακτική όλων των εργαλείων που έχουμε αναπτύξει, γιατί έχουμε στο παρελθόν αναπτύξει διάφορα εργαλεία, διάφορα μέσα στην τελευταία δεκαετία που δεν συνεργάζονταν μεταξύ τους. Έτσι πρέπει να μείνουν τα πράγματα. Πρέπει να πούμε ότι ε, τα στοιχεία που καταχωρίζω σε μια βάση δεδομένων ενός κράτους μέλους δεν θα επικοινωνούν με αυτά που καταχωρίστηκαν στην βάση δεδομένων ενός άλλου κράτους μέλους. Πρέπει να προχωρήσουμε και αυτό, όχι μόνο λόγω της κρίσης της, το μεταναστευτικού ή για οποιοδήποτε λόγο, αλλά και γιατί έχουμε τα μέσα και τις δυνατότητες. Και πάντα βέβαια αυτό ε, σε σεβασμό των κανόνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα, θα θυμάστε την εποχή που εγώ διαπραγματευόμουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν ε, ε, θεωρείται δεδομένο ότι το ένα θα κατά ε, τα άλλα. Και βεβαίως Συμβούλιο Κοινοβούλιο και ο ρόλος μας. Αυτό είπα και από την αρχή. Θέλω να αγωνιστώ Θέλω να ακούσω τις δικές σας τις θέσεις. Θέλω σε εσά να βρω το όργανο, το θεσμικό όργανο με το οποίο θα συνεργαστούμε, με το οποίο και θα βρούμε τις καταλληλότερες λύσεις σε σχέση με το Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και το Συμβούλιο. Υπάρχουν κρατημέλη που συμφωνούν με τα όσα είπατε και εσείς. Ρόλος μου λοιπόν είναι σε συνεργασία μαζί σας να ανεβρώ τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα χτίσουν ένα δρόμο συνεργασίας για να εξασφαλίσουμε τις λύσεις σε αυτή τη δέσμη. Όχι συμβιβαστικά, γιατί δεν είπα ότι θα συμβιβαστώ ποτέ στο πακέτο και τις προτάσεις που θα καταθέσουμε. Τελικά σχόλια για τις ημερομηνίε για το χρονοδιάγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προβλέπεται για τα τέλη Ιουνίου ε, τυπικά για να κατατεθεί κάτι, για να συζητήσει κάτι μάλλον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρέπει τρεις-τέσσερις εβδομάδες πιο πριν να έχει κατατεθεί το σχέδιο συμπερασμάτων. Έτσι λοιπόν, ω προ το χρόνο τουλάχιστον και το τυπικό, δεν μα εμποδίζει τίποτε να προχωρήσουμε τη δουλειά μα μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, εγώ λέω ότι ο σχεδιασμό μα μας επιβάλλει και κάποιε καταληπτικέ προθεσμίε. Για να είμαστε βέβαιοι ότι για το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι. Όλα αυτά θα πάνε κομμάτι-κομμάτι να μπουν στην ε, γραμμή και στο υλικό το οποίο περνώντας και από το Κορεπέρ θα μας οδηγήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και βεβαίως θα δείτε κι εσείς τι θα προκύψει ως αποτέλεσμα. Μίλησε ήδη για τους ε, ελέγχους στα ιστορικά σύνορα. Ε, και τα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα δείτε αν κοιτάξετε προσεκτικά τις προτάσεις ότι έχουμε κάνει ε, εκτεταμένη δουλειά για τη διαμόρφωση του που όχι μόνο στους τομείς που μας ενδιαφέρουν εδώ, που αναφέρομαι εδώ, ε, διαχείριση συνόρων, άμυφ και τα λοιπά εργαλεία ή ταμεία. Ε, υπάρχει πολλή δουλειά με προβολή αναγκών του μέλλοντος σε σχέση με τα όσα έχουμε δει να συμβαίνουν στο παρελθόν. Και έτσι στις 2 Μαΐου θα δείτε όχι μόνο τις γενικές αρχές του Πουδουπού, αλλά και τις συγκεκριμένες τομεακές δικές μας προτάσεις, θα τις δείτε κάπου στις αρχές ή μέχρι τις 12 Ιουνίου. Με αυτά, Πρόεδρε, ελπίζω να μην σας καθυστέρησα πολύ. Ε, διαβεβαιώνω και άλλη μια φορά την διθεσιμότητά μου για συνεργασία και συζήτηση όποτε το ζητήσετε. Βεβαίως και είστε ευπρόσδεκτοι και στις συνεδριάσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλή η πρώτη σας παρουσία εδώ. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, για την ε, αυτοπιθαρχία που επέδειξαν. Ας δούμε τώρα τι έχει να πει η Τάνια για τον τριμερή διάλογο και τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό. Τάνια. Είμαι... Ε, νομίζω ότι κατανοώ ότι δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω τώρα για το πού βρισκόμαστε στα πλαίσια του τριγωνικού διαλόγου για τον συγκεκριμένο κανονισμό. Καταρχάς, οι προϋποθέσεις για τη διεθνή προστασία είναι ένα από τα επτά κομμάτια της ισχύουσας νομοθεσίας για το άσυλο. Για τη διεθνή προστασία αναφερόμαστε ε, στο δύο σταδίων σύστημα το οποίο θεωρητικά ισχύει σήμερα στην Ευρώπη, γιατί στην ουσία οι πρακτικές είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια οδηγία η οποία συμπεριελήφθη αρχικά στην πρόταση του 2016 για την αναθεώρηση της χορήγησης ασύλου. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις το μήνα Σεπτέμβριο υπό την Προεδρία της Μάλτας. Είχαμε 14 συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο προσωπικού τεχνικού και ευχαριστώ όλους τους συμβούλους για την εξαιρετική βοήθεια και την ε, ε, Βουλγαρική Προεδρία. Επίσης είχαμε συνάντηση στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, προχώρησαν αρκετά τα πράγματα, αρκετά τεχνικά θέματα καταφέραμε να τα κλείσουμε. Κάποιες εκκρεμότητες παραμένουν, αλλά βασικός στόχος είναι να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε ε, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές να υπενθυμίσω ότι εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε μια ξεκάθαρη εντολή να γυτνιάσουμε και ε, την επικουρική προστασία ε, και την διαδικασία χορήγησης πενταετούς άδεια παραμονής έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις και τα επιπλέον κόστη. Αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία ακολουθούμε οι διαπραγματεύσει είναι δύσκολες, αλλά ελπίζω πριν από το καλοκαίρι να ολοκληρωθούν. Ευχαριστώ Τάνια. 16 Μαΐου είναι ο επόμενος ε, το ηγονικός διάλογος. Λοιπόν, συνάδελφοι, θα αρχίσουμε την ψηφοφορία στις 11. 11 να είστε όλοι εδώ με τις κάρτες σας. Θα ξεκινήσουμε, ελπίζω, εγκαίρως.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 Παρακαλώ καθίστε, πρέπει να ξεκινήσουμε. Um, I'm going to begin the vote. Um, I'm not sure about everyone else. Εγώ είμαι έτοιμος, εσείς δεν νομίζω. Colleagues, take your seats. Okay, we begin the vote uh, with... Uh... Ξεκινάμε με το σημείο 6, ετήσια έκθεση για τη λειτουργία της, του Σέγγεν, της ζώνης Σέγγεν εισηγητής ο κύριος Κοέλιο. Θέλετε το λόγο πριν την ψηφοφορία κύριε Κοέλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, μια μικρή εισαγωγή να χαιρετήσω την εξαιρετική συνεργασία με τους Κιώδης και να υπογραμμίσω ότι εμείς θα ψηφίσουμε την πρώτη κοινοβουλευτική έκθεση για το χώρο Σέγγεν. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα όχι μόνο για να προστατεύσουμε τους πολίτες και την ελευθερία διακίνησής τους, αλλά επίσης να διασφαλίσουμε τον δημοκρατικό έλεγχο από πλευράς του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Κοέλιο για την προσπάθεια την οποία κάνατε. Υπάρχει μια διόρθωση τεχνική της τελευταίας στιγμής. Στη σελίδα 6, το 84 δεν καλύπτεται στη συμβιβαστική 5α, αλλά στη συμβιβαστική 5. Στην περίπτωση δηλαδή που γίνει δεκτή, ε, τότε θα πρέπει η 84 ε, να ψηφιστεί ε, από μόνη της. Λοιπόν, περνάμε στις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε με τη συμβιβαστική παρήθμου 1. Ψηφίζεται. Άρχεται, ψηφίζεται. Κοιτάξτε, ετοιμαστείτε όλοι. Εξακολουθείτε να μπορείτε να ψηφίζετε πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή, συμβιβαστική 2, ψηφίζεται. Κύριε Πρόεδρε. Έρχεται η κάρτα μου, οπότε προς το παρόν θα ήθελα να ψηφίζω Ανατάσεως. Ή με το δάχτυλο, αν θέλετε, για να καταλαβαίνω. Συμβιβαστική 2 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Συμβιβαστική 10 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. 44 ψηφίζεται. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 3 ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 3α κεφαλαίο ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή συμβιβαστική 4 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Ο 78 ψηφίζεται. Τέλος. δεκτή ή μάλλον απερίφθει. Συμβιβαστική 5 ψηφίζεται. Συμβιβαστική 5 πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή. Συμβιβαστική 5α μικρό. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 6 ψηφίζεται. Τέλος. Συμβιβαστική 7 ψηφίζεται. Τέλος. Συμβιβαστική 16 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 101 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 24 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 103 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφη. Συμβιβαστική 32 ψηφίζεται. Τέλος. Κοιτάξτε, έχουμε ένα θέμα. Οι σοσιαλιστές έχουν ένα μέλος επιπλέον που ψηφίζει. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας, δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ, τέλος μάλλον. Συμβιβαστική 11α μικρό ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή 16α ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική. Α, συγγνώμη. Τροπολογία 115. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική 9. Ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 11 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 12 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 13 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 14 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 15 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 169 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 170 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 172 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική, α, λάθος, 174 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφη. Συμβιβαστική 26 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 177 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 178 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 17 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 186 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 18α μικρό ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 188 α, διορθώνει ο πρόεδρος. 187 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Συμβιβαστική 18 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 194 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 19 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 20α ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 20 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 20 β ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 21 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 22 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 22 β ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 221 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 22α ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 23 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 226 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 233 ψηφίζεται. Τέλος, δεκτή. 24α ψηφίζεται. Τέλος, δεκτή. 238 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 240 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 25 ψηφίζεται. ...247 ψηφίζεται. Τέλος. ...249 ψηφίζεται. Τέλος. απερίφη Τώρα περνάμε στην 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή. 2. Τέλος. Δεκτή. 3. Τέλος. Δεκτή. Τέσσερα. Τέλος. Δεκτή. 27 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 28 υπέρ. Ε, Τέλος. Δεκτή. 28α ψηφίζεται. Α, για μια στιγμή. Τέλος. Δεκτή. 28α ψηφίζεται. Συγγνώμη, μόλις το κάναμε αυτό. Έκανα λάθος. 18 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 29 ψηφίζεται. Τέλος. Η 22 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 30 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. 32 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Συμβιβαστική 31 ψηφίζεται. Τέλος. Δεκτή. Τριάντα οκτώ ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Τριάντα εννέα ψηφίζεται. Τέλος. απερίφθη. Σαράντα ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Ονομαστική κλίση ψηφίζεται για το σύνολο. Τέλος. 45 υπέρ 8 κατά 3 αποχές συγχαρητήρια στον κύριο Κοέλιο. Καλώς. Λοιπόν, κράτησε πολύ ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα Λοιπόν, παρακαλώ ησυχία. Λοιπόν, έκθεση Φεράρα. Ησυχία παρακαλώ. Έχετε λάβει τον τελικό κατάλογο ψηφοφοριών και ένα κείμενο με τις τελικές ψηφοφορίες και ένα κείμενο με εναλλακτικέ ε, διατυπώσεις για τις ε, συμβαστικές 42, 43, 44 και αν δεν εγκριθεί η συμβαστική 39. Αυτό, όλα αυτά θα χρειαστεί να τα δούμε αν δεν εγκριθεί η συμβαστική 39. Λοιπόν, τι θα ψηφίσουμε. Κοινή διαδικασία για διεθνή προστασία στην Ένωση. Η συγκήτρια η Λόρα Φεράρα θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους όλους <clears throat> για την εξαιρετική συνεργασία ήταν δύσκολη δουλειά. Ξεκινήσαμε από τον Οκτώβριο του 2016. Ένα μισή χρόνο δηλαδή δουλέψαμε. Εντατικά. Και γιατί ήταν τεχνικός ο χαρακτήρας του κανονισμού, αλλά και γιατί ήταν λεπτά πολιτικά τα ζητήματα. Νομίζω ότι με το τελικό κείμενο μπορούμε να πούμε ότι πραγματοποιούμε ένα βήμα προόδου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ασύλου με όλα τα στοιχεία αυτά που θα χρειαστούν ε, να τις συμπληρώσουν ώστε να έχει μια ταχεία αποτελεσματική διαδικασία αλλά πάνω απ' όλα ενιαία διαδικασία για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ τους και ηγητές που με συνόδευσαν, μου παραστάθηκαν σε αυτή τη διαδικασία αλλά και όλο το προσωπικό που μας ε, προσέφερε την αρρωγή του. Ευχαριστώ. And Ναι, όπως είπα για την έκθεση Κοέλιο, όταν ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης, δεν το κάνω για λόγους τυπικής ευγένειας. Ξέρω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ δύσκολο και ότι όλοι εργάστηκαν πολύ. 188, 189 ε, τροπολογίες ε, από κοινού. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. 188 και 189 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. απορρίπτονται. 190. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 191 και 192 ταυτόσιμες άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Στα α τώρα. 477. Άρχεται. Πέρας. απολύπτεται Ωραία. Τροπολογία 33 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία ε, 480. Άρχεται. Α, καταπίπτει. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, μισό λεπτό. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι είχε δίκιο ο πρόεδρος ε, και άδικο η γραμματεία. Έτσι νομίζω πείθεστε ότι ελέγχω την κατάσταση. Ψηφίζουμε την 480. Άρχεται. 480. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 485. Άρχεται. Πέρας. 485. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται. Συμβαστική 1. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 στο άρθρο 5 άρχεται. Συμβαστική 2 για το άρθρο 5 άρχεται. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 για το άρθρο 6 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5.65 άρχεται. 5.65. Α, όχι. Συγγνώμη, καταπίπτει. Καταπίπτει λέμε. Συμβαστική 4α. 4α. Αντί να βρει, συγγνώμη, δικό μου λάθο. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Συμβαστική 6. Στη σελίδα 15, αν έχετε τον ίδιο κατάλογο ψηφοφορίων όπως και εγώ, Άρχεται. Συμβαστική 6. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Στη σελίδα 17 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαστική 11 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαστική 12 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 7.96. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 7.97 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 7.99 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 7.98 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 800 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 801 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Οκτακόσια δύο, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 874. Άρχεται. 874. Πέρας. Απορρίπτεται. 875. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 8.78 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 8.77 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 8.76 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 880. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 881. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 882. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Το συμβαστική 19 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 926. Άρχεται. 926. Άρχεται πέρας. Εγκρίνεται. 927. Εγκρίθηκε. Εντάξει, παρακολουθείτε όλοι. Λοιπόν, πού ήμασταν, 9.27. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22α. Άρχεται. Πέρας. Συμβαστική 23. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Στη σελίδα 52 συμβαστική 26 άρχεται. 26 συμβαστική σελίδα 52. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 30. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεβαστική 31. Άρχεται. Στη σελίδα 60 είμαστε. Άρχεται είπαμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1174. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Άρχεται. Πέρας. Αγκρίνεται. Συμβαστική 33. Άρχεται. Συμβαστική 33. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 35. σύνταξη 63. Ή συμβαστική Α, συγγνώμη, όχι, Α, συγγνώμη. Α, πήδηξα μια σελίδα. Δεν θα ήταν σωστό αυτό. Λοιπόν, τροπολογία 12.47 στη σελίδα 70 άρχεται. 12.47 στη σελίδα 70 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 12.53 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα, συμβαστική 35 στη σελίδα 73 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 36 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 37. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 38 στη σελίδα 79. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα Στη σελίδα 83, η τροπολογία 1398 άρχεται. 1398 άρχεται πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 39 άρχεται. Συμβαστική 39. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Συμβαστική 40. 40 άρχεται. Συμβαστική 40. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 41 άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 42. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 43. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 44. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τροπολογία 1502. 1502 στη σελίδα 90 άρχεται. Όχι, 1502. Και 1503 γιατί είναι ταυτόσιμες, ναι. Εντάξει. Τις ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. 15.04. Άρχεται. 15.04. Πέρασε. Εγκρίνεται. 15.06. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 15.07. Όχι, συγγνώμη. 15.08. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, Δικό μου λάθος, δικό μου λάθος. Μπορούμε να ψηφίσουμε τη 15, πρέπει να ψηφίσουμε τη 15.07. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Εντάξει, πέρας. Εγκρίνεται. Το 1509 άρχεται πέρας. Δεκαπέντε δέκα. συγγνωμη Συγγνώμη, ε, ξέρετε ότι αυτή η ψηφοφορία έχει κρατήσει πολλή ώρα. Πέρας για 15-10. <clears throat> Εγκρίνεται. Συμβαστική 45. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 46 στη σελίδα 94. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 47. Στη σελίδα 96 άρχεται. Συμβαστική 47 έλεγα. Πέρασε. Εγκρίνεται.

Συμβαστική 48 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 1584 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, περνάμε στη 1590. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 1592. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 1595 και 1596 ταυτόσιμες άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται. Λοιπόν, οι ε, σκέψεις τώρα. 195. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 196. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 197 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 199 άρχεται. 199 πέρας. Απορρίπτεται. 201 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 203 άρχεται πέρας. Εγκρίνεται. 204 άρχεται πέρας. Απορρίπτεται. 207 άρχεται πέρας εγκρίνεται. 209 άρχεται πέρας απορρίπτεται 215 2.15. Πέρας. Απερίφθη. 2.16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Διακόσια σελίδα 132 και 258. Όχι, όχι, δεν είναι ο λάθος. 257 και 4, τέλος πάντων, έχετε ήδη ψηφίσει. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα την ψηφοφορία, τώρα την κλείνουμε. Απερίφθη. Σαν. 258. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 264. Αρχίζει. Πέρασε. Εγκρίνεται 273. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται 284, άρχεται. Πέρας. Απερίφθη 285, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται υπαριθμόν 7, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 296 τώρα, άρχεται. Πέρας. Απεριφθεί. Υπαριθμόν 9. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 301. Άρχεται. Πέρας. Και απεριφθεί. Τρακόσια τριάντα εννιά. Σελίδα οχτώ, Άρχεται. Πέρας. Απεριφθεί. 340 άρχεται Πέρας. Και εγκρίνεται. 344. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 342. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 341. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 403 είναι. Λέει ο πρόεδρος. 423. So we go to the end now? No, there's page 115. Yeah. So sorry for the Με συγχωρείτε για την ε, μικρή διακοπή, αλλά ήθελα να είμαι βεβαίω ότι θα κάνουμε λάθος. 403 τώρα, στη σελίδα 115. 423. Αν έχει κάποιο άλλο αντίρρηση, παρακαλώ να μου το επισημάνετε να το εξετάσουμε, αλλά αν δεν κάνω λάθο, έχουμε πάει στο 423. 423 στη σελίδα 115. Έχει καταπέσει και αυτή. 423. 423 αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι η σωστή τροπολογία. Ξέρω ότι δεν έχει πολύ κύρος η φωνή μου, αλλά παρακαλώ βοηθήστε να ψηφίσουμε τα 423. 423, εκτός και αν έχει κάποιος αντίρρηση να το συζητήσουμε. Συντονιστής του ΕΛΚΑ. 422 και 423 για το δικό μας κατάλογο ψηφοφοριών ε, σημειώνονται ως ταυτόσιμες. Όχι, όχι, είναι χωριστά 423 λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, έχει δίκιο να πληρωτήσει συντονιστής του τον και τον ευχαριστώ. Καλά έκανα και ζήτησα τη γνώμη σα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε περάσει ήδη στην 426 με αυτή την επιχειρηματολογία. Όλα τα άλλα έχουν καταπέσει και πάμε στην 426. Ευχαριστώ πάλι για την βοήθεια. Ψηφίζουμε 426, έτσι δεν είναι. Θα επαληθεύσω. Αν έχουμε 426 να ψηφίσουμε για να προχωρήσουμε προς το τέλος. Αγαπητοί συνάδελφοι, σα σας προτείνω το εξής. Μπορούμε να πάμε στην τελική ψηφοφορία, αλλά προτείνω να ψηφίσουμε από την 30 και μετά. Θα είναι καλύτερα και πιο απλά τα πράγματα για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Από την 30 και μετά ψηφίζουμε λοιπόν. Όχι. and 56 were adopted. Επειδή έχουν εγκριθεί οι 1595 και 1596. Because 1595 and 1596 were adopted. Επειδή έχουν εγκριθεί 1595 και 1596, οι 30 και οι 42 δεν καταπίπτουν και άρα πρέπει να ψηφιστούν. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. 30 και 42 που είναι ταυτόσιμες. Ναι, όντως. 4.22. Ετιολογική σκέψη 62 με την τροπολογία 30 και την 4, 22. άρχεται, πέρας, σελίδα 114. Εγκρίνονται. Τώρα στην 426 άρχεται. 426. Πέρας. Απερίφθη. 31 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται.

Πέρας. Απερίφθη 443. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 454 στη σελίδα 117. Άρχεται. Πέρας. Απεριφθεί. 454. Κυρία Νετσφέλτ. Ε, μπορούμε να ξαναδούμε αυτή τη ψηφοφορία, γιατί δεν είχαμε καταλάβει τι ψηφίζουμε, τουλάχιστον εγώ. Να το ξανακάνουμε. 454 στην αιτιολογική σκέψη 75, έτσι. Ναι, λέει ο πρόεδρο, αλλά αν δεν ήταν σαφέ. Α επαναλάβουμε την ψηφοφορία. 454, ξανακάνουμε την ψηφοφορία. 454, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 455, άρχεται. Πέρας.

Απερίφθε. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστικά παρακαλώ. Ξεκινάμε. Has everyone voted? The votes. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. 36 υπέρ 12 κατά 8 αποχές και συγχαρητήρια στην κυρία Φεράρα. Ναι, συγγνώμη και η εντολή για την ανάληψη των ε, συνομιλιών, των διαπραγματεύσεων. Ψηφίζουμε τώρα πάλι ηλεκτρονικά. Πέρας. Και εγκρίνεται 39 υπέρ 9 κατά 4 εποχές. χαρακτήρια κυρία Φεράρα και σε όλους τους σκιώδες που συνεργάστηκαν στην υπόθεση αυτή. Colleagues, we have a further two. Colleagues, okay, colleagues, we go straight to the next votes. Περνώ απευθείας στις επόμενες προφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώντας σας για την υπομονή σας. Έτιας, Με την κυρία Γκάλ την οποία και ρωτώ αν θέλει να λάβει το λόγο. Πολύ στο... Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω μόνο να σας ενημερώσω ότι το Κορεπέριο θέτησε τις θέσεις του Κοινοβουλίου μετά τις τελευταίες τεχνικές επαφές. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία της δύο προεδρίες, ε, ιδιαίτερα τη βουλγαρική. Πάντως πρέπει να ξέρετε ότι ήταν πολύ περίπλοκο το θέμα. Κάναμε πολλά. Έχουμε μια σαφέστατη θέση του Κοινοβουλίου που βεβαιώνεται και από το κείμενο και προς τους κοιόδης, την κυρία Γκίωμ, τον κύριο Ντεπρέ, την κυρία Στέβεν, την κυρία Βερζιά και τους λοιπούς. Θέλω να πω ότι μπορεί να είχαμε μερικές φορές έντονες αντιπαραθέσεις, αλλά πάντως αυτές βοήθησαν και συνέβαλαν στην ε, διαμόρφωση ενός καλού κειμένου, ενό σαφού κειμένου που μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη. Και πάνω απ' όλα θέλω να, να, βοηθ, να ευχαριστήσω του ε, βοηθού ε, πολιτικού συμβούλου των πολιτικών ομάδων που έκαναν εξαιρετική δουλειά. Με πολλή υπομονή για να εξετάσουν όλα τα τεχνικά ζητήματα. Ιδιαιτέρως πρέπει να ευχαριστήσω δε, τη γραμματεία μας και την Κατρίν Χιούμπεν για αυτή την εξαιρετική δουλειά που έκανε, έπρεπε ρητά να αναφέρω το όνομά της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κίνγκα και ιδιαίτερα για τη ρητή αναφορά στις προσπάθειες και το έργο της γραμματείας και του προσωπικού μας, πράγμα από το οποίο δεν γίνεται συχνά. Προχωρώ λοιπόν. Πρέπει να αναφέρω τη διαδικασία. Λοιπόν, πρώτη διαδικασία. Εάν εγκριθεί. Όχι. Πάμε στην ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Απλώς ήθελα να επενέσω την γραμματεία μας. Εν πάση περιπτώσει. Πέρασε. Και εγκρίνεται με 45 υπέρ, 10 κατά, 0 αποχές. Η δεύτερη ψηφοφορία. Αρχίζουμε. Πέρας. Α, κυρία Βεργιά, για μετά είσαστε εσείς μάλιστα. Ευχαριστώ που μας διευκολύνετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Μα δεν εμφανίστηκε ο οθόνες. Εγώ τουλάχιστον στη δική μου οθόνη δεν είδα το αποτέλεσμα. Μου είπαν όμως ότι είναι 45 υπέρ 10 κατά 0 αποχές. Γιατί δεν εμφανίστηκε στην οθόνη. Δεν εμφανίστηκε σε όλες τις οθόνες από ό,τι μου λένε. Παράξενο κάπως. Μπορεί αυτό να είναι πρόβλημα, όχι, γιατί έχετε κάνει την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Okay, fine. Okay, I don't want to create some problems, but that's the... Όχι, όχι, δεν θέλω εγώ να κολλήσει εργό, αλλά φοβόμουν πως οδηγούσε σε κάποια προβλήματα το ότι δεν εμφανίστηκε το αποτέλεσμα. 45 υπέρ 10 κατά 0 αποχές και στη δεύτερη και συγχαρητήρια στην κυρία Γκάλ και στους Σκιώδης. Κυρία Βερσιά, δικαστικό εσείς. Ναι, Πρόεδρε, και επί τη ευκαιρία θα ευχαριστήσω και εγώ, όπως και η Κίνγκα, όλους τους συνεργάτες μας, αλλά έχω μια παρατήρηση στον τρόπο με τον οποίο χρειάστηκε να εργαστούμε. Σταματήσαμε τις συζητήσεις των σκιωδών ε, το τέλη Δεκεμβρίου υπό την Εστονική Προεδρία. Πέρασαν τρεις μήνες και με λεγόμενες τεχνικές συζητήσεις όπου κάποια στιγμή ήρθε και μια συνενετική, μια συμβαστική πρόταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που με τα βία τα προστατεύει. Καθόλου ικανοποιητικό όλο αυτό και γι' αυτό και τι ευχαριστώ πολύ το προσωπικό. Παρακαλώ στο μέλλον να μην ακολουθηθούν αυτές οι μέθοδοι που δεν είναι χρήσιμες για κείμενα τόσο σημαντικά και νομοθετικά γιατί ε, θα υπαγάγουν υπηκόους τρίτων κρατών που δεν χρειάζονται ε, προξενική θεώρηση στην υποχρέωση για την λήψη άδεια ταξιδίου. Επιβάρυνση περιττή. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό και δεν έπρεπε να ε, περάσουμε από αυτή τη διαδικασία. Επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους μεθοδολογή, μέθοδοι εργασίας δεν είναι καλές. Στο πόδι. Ενώ ήταν τόσο σημαντικό το κείμενο μπορούσαμε να δώσουμε και μερικές εβδομάδες δουλειάς παραπάνω για να το κάνουμε καλό. Ο πρόεδρος δεν ήταν και διαδικαστικό, κυρία Βεργιέ. Σχόλιο ήταν. Νομίζω ότι τα άκουσα τα σχόλιά σας η συγκήτρια, όπως και οι λοιποί συνάδελφοι, αλλά δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση. Πάτε στο είπατε ότι είχατε να πείτε. Um, Καλώς συναδελφοί, θα πάμε στο σημείο 10. Και ο Τζουέξλερ είναι μαζί μας. Είναι το τελευταίο σημείο για σήμερα το πρωί, το σημείο 10 Okay, as he comes uh, to the front, this is a presentation by the legal service. Some of you be following this uh, judgment. Λοιπόν, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της 22ης Μαρτίου 2018 στην υπόθεση Καπιτάνη, καπιτάνη-δεκαπιτάνη ε, εις βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. σχετικά και με τον τριμερή διάλογο και τις ε, συνεχιζόμενες νομοθετικές διαδικασίες και τις συνέπειες που έχει αυτή η απόφαση. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας για να μας παρουσιάσει λεπτομερώς την γνωμοδότησή του και μετά μπορεί να ακολουθήσει μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Ο κύριος λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μας δίδεται να παρουσιάσουμε ε, την υπόθεση αυτή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Είναι η πρώτη φορά που, ένα γενικό, που το Γενικό Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ασχολείται με την υπόθεση αυτή σχετική με μια νομοθετική ε, πρωτοβουλία, διαδικασία και με τους τριμερείς διαλόγους και τις τετράστιλες ε, σελίδες των εγγράφων. Εξετάστηκε από το 7ο Σώμα του Δικαστηρίου. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση Πολλοί πιστεύουν ότι είναι σταυροδρόμη η απόφαση αυτή με πολύ συγκεκριμένες συνέπειες οι οποίες ξεπερνούν την απλή πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα. Θεωρητικά βέβαια περί αυτού πρόκειται πρόσβαση του κοινού στα νομοθετικά έγγραφα. Κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αίτημα το οποίο κατέθεσε ο Εμίλιο Ντεκαπιτάνη για πρόσβαση σε έγγραφα. Ο κύριος Ντεκαπιτάνη αρχικά παρουσίασε ε, ένα ευρύτατο αίτημα που κάλυπτε το σύνολο σχεδόν των εγγράφων, συγκεντρώνοντας την προσοχή του στα έγγραφα των τεσσάρων ε, με τις τέσσερις στήλε για τις ε, ενεξελίξει νομοθετικές διαδικασίες. Το αίτημα αυτό ε, σε μια δεύτερη φάση περιορίστηκε από τον ίδιο τον κύριο Ντεκαπιτάνη στις, ε, στις τρέχουσες διαδικασίες με βάση τον τίτλο 5 της Συνθήκης σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες στον τομέα των ελευθεριών δικαιοσύνης εσωτερικών υποθέσεων, όπως επίσης και με βάση το άρθρο 16. Το Κοινοβούλιο ενημέρωσε τον ετούμενο ότι έχει εντοπίσει 7 τετράστιλα τέτοια έγγραφα και του έδωσε πλήρη πρόσβαση σε 5 και επιμέρους πρόσβαση σε 2. Αυτό σημαίνει ότι στα δύο αυτά έγγραφα η τέταρτη στήλη δεν διετέθη. Είναι προτάσεις άλλωστε με τις οποίες ασχολήθηκε και η δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον κανονισμό Europol. Τα επιχειρήματα λοιπόν τα οποία έγιναν, τα οποία ε, ακούστηκαν μάλλον, καλύπτουν δύο επίπεδα θα έλεγα σκέψεων, δηλαδή συγκεκριμένες παρατηρήσεις σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση και το θέμα που συζητήθηκε ήταν η ευαισθησία της συζήτησης αυτής και υπήρξαν και κάποιες γενικότερες συζητήσεις σχετικά με τη λειτουργία της νομοθετικής διαδικασίας. Ο κύριος Ντεκαπιτάνη αμφισβήτησε ε, στο δικαστήριο λοιπόν την στάση του Κοινοβουλίου, παρενέβη ε, το Συμβούλιο, παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζοντας το Κοινοβούλιο και στο τέλος Μαρτίου το δικαστήριο αποφάσισε, πήρε την τελική του απόφαση. Σχετικά τώρα με την απόφαση αυτή πρέπει να πούμε ότι καταρχάς το δικαστήριο λέει ότι η νομολογία και όλες οι αποφάσεις οι σχετικές με, με τον κανονισμό 1049 2001 ε, ε, περιγράφουν την φύση των τριμερών ή τριγωνικών διαλόγων και η απόφαση επίσης ε, χρησιμοποιεί και επιμέρους επιχειρήματα και ασχολήθηκε πρώτα με την γενική προϋπόθεση μη πρόσβασης. Ε, θεωρούσαμε ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να θεωρήσει δεδομένη την μη πρόσβαση στην τέταρτη στήλη στον βαθμό που οι διαδικασίες νομοθετικού τύπου είναι ανοιχτές, είναι ε, τρέχουσες. Όμως το δικαστήριο δεν δέχθηκε την ιδέα αυτή ε, γιατί στηρίχθηκε στο επιχείρημα ότι μια τέτοια αντίληψη είναι κάτι το οποίο δεν είναι αντίθετο με την εύρυθμη νομοθετική διαδικασία. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν η απόφαση ε, σέβεται πλήρως την απόφαση Τούκο ε, και άλλη μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και τέλος το δικαστήριο συνέχισε και μπήκε στην ουσία και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ασχολήθηκε λοιπόν με τον κίνδυνο υπονόμευσης της νομοθετικής διαδικασίας μέσω αυτού του τύπου ενημέρωσης και κάνοντας αυτό ακολούθησε την απόφαση την οποία είχε λάβει το ίδιο το Κοινοβούλιο ε, η απόφαση αναφέρεται λοιπόν στην αιτιολόγηση της ε, υπόθεσης της ευαισθησίας του θέματος στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας, κάτι το οποίο ήταν ε, το αντικείμενο της πρότασης και απέρριψε την αντίληψη αυτή. Λέγει ότι ακόμα και αν το θέμα είναι νομικά και πολιτικά δύσκολο, η ευαισθησία του λεγόμενου αστυνομικού τομέα δεν μπορεί να αποτελέσει ένα επιχείρημα το οποίο να υπονομεύσει την πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα. Αυτά περιλαμβάνονται στα σημεία 89 με 97. Και δεύτερον, το Γενικό λοιπόν, Δικαστήριο, το Δικαστήριο Γενικών Υποθέσεων ασχολήθηκε με τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπολείπων οργάνων γενικότερα για τα θέματα των νομοθετικών διαδικασιών. Εδώ το πρώτο επιχείρημα είναι ότι ο κίνδυνος ε, της δημόσιας πίεσης προς τους ε, ασκούντες αυτήν την διαδικασία, εδώ το δικαστήριο λέγει ότι η έκφραση της κοινή γνώμης είναι αναπόσπαστο τμήμα της άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι λοιπόν προσθέτει το δικαστήριο ότι ακόμα και αν η πίεση αυτή της κοινή γνώμης θα μπορούσε να αποτελέσει επιχείρημα αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης άρνησης πρόσβησης, πρόσβασης, το δικαστήριο αναγνωρίζει με βάση και την προηγούμενη νομολογία ότι η πραγματικότητα μιας τέτοιας πίεσης θα πρέπει να γίνει αντιληπτή με ε, βεβαιότητα και να ε, χρησιμοποιηθούν και να παρουσιαστούν απτές αποδείξεις για το αρνητικό της πίεσης αυτής. Κάτι το οποίο δεν συνέβη, ως εκ τούτου το επιχείρημα του Κοινοβουλίου απορρίπτεται. Τώρα, ε, το επιχείρημα του προσωρινού και ενδιάμεσου χαρακτήρα του εγγράφου και εδώ το δικαστήριο απέρριψε το έγγραφο αυτό λέγοντας ότι στην εξαίρεση που είχε χορηγηθεί στα πλαίσια της απόφασης 1049 δεν περιλαμβάνεται ή δεν σημειούται η αδίποτε διάκριση σχετικά με το έγγραφο, αν είναι προσβάσιμο σε διαφορετικές φάσεις ε, των, ε, της νομοθετικής διαδικασίας. Επίσης, το επιχείρημα ε, σταδιακής απώλειας εμπιστοσύνης ανάμεσα στα όργανα. Εδώ χρησιμοποιήθηκε το αντεπιχείρημα του καθήκοντος συνεργασίας των ε, εκπροσώπων των νομικών. Εάν υπήρχε απώλεια εμπιστοσύνης ανάμεσα στα όργανα, τα όργανα θα έπρεπε να, ε, τότε σε αυτή την περίπτωση θα παραβίαζαν το καθήκον τους για θεμητές μορφές ε, συνεργασίας. Συνεπώς λοιπόν ο κίνδυνος για την απώλεια εμπιστοσύνης ανάμεσα στα όργανα δεν τεκμηριώθηκε. Και στο τέλος ένα γενικότερο επιχείρημα του Κοινοβουλίου, το οποίο απερίφθη, λέγοντας ότι οι τριμερείς διάλογοι, και ξεκαθαρίζεται αυτό, είναι ουσιαστικό κομμάτι της νομοθετικής διαδικασίας ως έχουν σήμερα. Αυτό περιλαμβάνεται στο σημείο 105 στο πλαίσιο αυτό λοιπόν παρατηρείται επίσης ότι το Δικαστήριο Γενικών Υποθέσεων επέμεινε λέγοντας ότι η απόφαση αυτή δεν αναφέρεται αποκλειστικά στο θέμα της άμεσης πρόσβασης των εργασιών των τριμερών διαλόγων, αλλά στο αίτημα μετά, στο αίτημα μάλλον, στην υπόθεση ε, άμεσης πρόσβασης μετά από συγκεκριμένο αίτημα του συνόλου των εγγράφων. Επίσης ε, δεν αναγνώρισε την δυνατότητα συμμετοχής στο σύνολο των συζητήσεων ανάμεσα στα θεσμικά όργανα ε, γιατί πολλές φορές ε, η τέταρτη στήλη γίνεται αντικείμενο ακριβώς των συζητήσεων αυτών. Τώρα, το επιχείρημα της, του προσωρινού χαρακτήρα της άρνησης και αυτό απερίφθη, λέγοντας ότι η διάρκεια των τριμερών διαλόγων μπορεί να κρατήσει αρκετά σημαντική χρονική περίοδο και μάλιστα χρησιμοποιεί ε, το δικαστήριο την έκφραση ε, να μην υπάρχει προβλέψιμο πέρας της διαδικασίας. Τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται ας πούμε σε επιτροπές του Κοινοβουλίου και τα οποία λαμβάνονται εσωτερικά σε σχέση με την συνέχιση και την ενημέρωση της, για την συνέχιση των διαλόγων είναι κάτι το οποίο δεν θέτει σε αμφισβήτηση την εμπιστευτικότητα της τέταρτης στήλη στο βαθμό ε, που συνεχίζεται ο τριμερής διάλογος. Λοιπόν, το Δικαστήριο Γενικών Υποθέσεων κατέληξε ότι κανένα από τα επιχειρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν επαρκές για να αποδείξει ότι η πρόσβαση στο έγγραφο τεσσάρων στυλών ή στα έγγραφα τεσσάρων στυλών θα μπορούσε να υπονομεύσει την νομοθετική διαδικασία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και γι' αυτό η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ακυρώθηκε και έτσι υποχρεούται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα έγγραφα. Τώρα, σχετικά τώρα με τις ε, πρακτικές συνέπειες αυτής της απόφασης. Σε σχετικά με μελλοντικά αιτήματα πρόσβασης σε αντίστοιχα έγγραφα, ε, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, ε, τότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εφαρμόσει ε, την απόφαση αυτή. Δεν μπορεί να θεωρήσει ότι είναι γενικευμένη η αντίληψη απαγόρευση στην πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή συνεχίζονται οι διαδικασίες. Τώρα, κατά περίπτωση, εάν θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης της διαδικασίας λήψεων αποφάσεων, αυτές αποδείξεις ε, προς, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Και τώρα σχετικά με τις γενικότερες συνέπειες, για τον τρόπο γενικότερης λειτουργίας των τριμερών διαλόγων δηλαδή, η απόφαση παραδέχεται ότι οι ε, τριμερής διάλογοι είναι τμήμα της νομοθετικής διαδικασίας και παραδέχεται επίσης ότι οι τριμερής διάλογοι ε, γίνονται, διεξάγονται και κλεισμένων των θυρών. Κατά τα άλλα όμως, οι περαιτέρω συνέπειες της έκδοσης αυτής της απόφασης για έγγραφα εκτός των εγγράφων τεσσάρων στυλών είναι δύσκολο στην παρούσα φάση να, ε, να υπολογιστεί το βάρος της απόφασης. Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι η απόφαση ελήφθη από το Δικαστήριο Γενικών Υποθέσεων είναι μια συλλογική διαδικασία. Έφεση μπορεί να υπάρξει μόνο με βάση την ομολογία και υπάρχει μια προθεσμία χρονική επίσης για την έφεση και η προθεσμία είναι η 8η Ιουνίου του 2018. Αυτά με λίγα λόγια μπορούμε να πούμε για την υπόθεση Δεκαπιτάνη. Είμαι στη διάθεσή σας. Ε, μπορεί να υπάρξουν ερωτήσει, αλλά έχουμε μόνο 10 λεπτά. Οπότε, η επόμενη φάση είναι η ενδεχόμενη ε, έφεση. Αυτό θα το εξετάσει βέβαια η Νομική Επιτροπή, αλλά για τα θέματα διαφάνεια η Επιτροπή μα είναι η κυριότερη. Υπάρχουν απόψει για το τι θα πούμε στη Τζούρι. Θα ήταν σημαντικό να τι ξέρουμε. The Young, η Σοφή. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Α, και η κυρία Ζίπελ. Ωραία, τρει. Ο κύριο το Ευχαριστώ. Ε, υπάρχει μια προσφυγή που, κάνει, ε, που έχω κάνει προς τον διαμεσολαβητή για την, πρόσφαση, για την πρόσβαση στο σε έγγραφα και περιμένω την απάντηση και για το μικρό διαφάνειας. Με θαρρύνει αυτή η απόφαση. Ελπίζω επιτέλους να υπάρξει λίγο περισσότερη διαφάνεια, να ανοίξει κάπως η στάση τους. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω επί της ουσίας. Και έχω και μια σύσταση για την διαδικαστική συνέχεια. Τι δεν καταλαβαίνω. Αυτό που λέγεται για την υπονόμευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εάν υπάρχει κίνδυνος εξωτερικής πίεσης. Και το δικαστήριο λέει ότι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να ασκήσουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα. Και θα πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση να μπορούν να παρακολουθούν την διαδικασία λήψη αποφάσεων. Εγώ νομίζω ότι σε μια δημοκρατία Γιατί αν κάποιο παρακολουθεί μια διαδικασία λήψη αποφάσεων, να μην μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του, αν είναι θέματα που τον αφορούν ή γενικότερα. Δεν νομίζω ότι αυτό υπονομεύει τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι κρύβεται πίσω από αυτό το επιχείρημα, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει κάποια διευκρίνηση. Και θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα κάναμε μεταξύ Είμαι ακόμη σκιώδης ενός θέματος που έχει κολλήσει στο Συμβούλιο. Είναι η πρόσβαση στα έγγραφα. Όπως ξέρει και η Σοφή, είχαμε υιοθετήσει πολύ καλή άποψη γι' αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να εξοπλίσουμε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου για να προχωρήσουν διαπραγματεύσει και αυτό το θέμα πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία. Δεύτερον, αντί να επιχειρήσουμε έφεση, καλά αυτό βέβαια θα το συζητήσει η νομική επιτροπή. Ω κοινοβούλιο δεν θα μπορούσαμε να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και σε περιπτώσεις ε, πολύ σαφείς όπως οι διαπραγματεύσει για το Μητρό Διαφάνειας. Ξέρω ότι οι πράσινοι ήδη ζήτησαν να δημοσιεύσουμε με δική μας πρωτοβουλία αυτό το έγγραφο τεσσάρων στυλών, το οποίο ακριβώς ε, είναι σύμφωνο και με το, την απόφαση του δικαστηρίου. Δηλαδή να μην περιμένουμε να μας κάνουν αίτηση, αλλά να δημοσιεύουμε αυτοβούλως εμείς αυτά τα κείμενα. Ευχαριστώ κύριε Τεγιόν. Η πρόσβαση στα κείμενα πρέπει να είναι το θέμα που έχει μπλοκάρει για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ουδέποτε. Του χρόνου εισηγητής μας δεν θα είναι πλέον εισηγητής. Τέλο πάντων, μπούμε σε αυτέ τι λεπτομέρειε. Και το θέμα τη μπλε κάρτα βεβαίω. Ε, ίσως και αυτό θα μπει στην ιστορία ω το θέμα με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση. Η Σοφή. Συμφωνώ με τον Ντένι Τεγιόν. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε έφεση. Ω κοινοβούλιο θα ήταν άθλιο. Θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την απόφαση. Για την λεγόμενη εξωτερική πίεση. Μα είναι το αντίθετο που ισχύει. Εξωτερικές πιέσεις προκύπτουν από τη μυστικότητα. Αν υπάρχει διαφάνεια, τι η πίεση. Εκτό βέβαια αν δεν έχει ε, σπονδυλική στήλη. Ραχοκοκαλιά, αλλά εκεί δεν θα σε βοηθήσει η μυστικότητα. Νομίζω ότι αν είναι μυστικέ διαπραγματεύσει μπορούν να σου ασκηθούν μεγαλύτερε πιέσει. Και δεύτερον, αν όντω ίσχυε ότι η γνωστοποίηση κειμένων θα υπονομεύσει συγκεκριμένα την νομοθετική διαδικασία, μα τότε πολλά κείμενα μπορείς να βρεις μέσω ΜΚΟ ή από το State Watch για όλα τα θέματα. Αν θέλεις, μπορείς να βρεις τα έγγραφα. Μόνο μια φορά δεν βρήκα ένα έγγραφο και ποτέ δεν υπονόμευσε αυτό την νομοθετική διαδικασία. Βλακώδες επιχείρημα. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα για το θέμα αυτό, στη συνέχεια θα πρέπει πραγματικά να χαιρετήσουμε αυτή την απόφαση και να κάνουμε αυτοβούλος ε, δημοσίευση. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ε, ευανάγνωστα αυτά τα κείμενα και ευχάριστα. Κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί τόσο πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρονται. Πιστεύω, λοιπόν, ότι όχι μόνο πρέπει να αναζωογονήσουμε αυτό το θέμα της, ε, του κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα, αλλά να έχουμε και αυτή την ετήσια έκθεση όπως κάνουμε παλιότερα για την πρόσβαση στα έγγραφα και την διαφάνεια. Επανειλημμένα το σώμα μας έχει πει ότι οι τριμερείς διάλογοι πρέπει να είναι πιο διαφανείς, τα έγγραφα να είναι πιο διαθέσιμα. Αλλά όταν το ψηφίσαμε φαίνεται ότι δεν καταλάβαμε τι ψηφίσαμε. Αλλά η Ένωση αλλάζει, το Κοινοβούλιο αλλάζει, πολύ περισσότεροι συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ένα χρόνο πριν τι ευρωεκλογέ να δείξουμε ότι ασχολούμεθα σοβαρά με τη διαφάνεια και είμαστε διαδεδομένοι να αλλάξουμε και τι δικέ μα διαδικασίε για να γίνουμε πιο ανοιχτοί. Ευχαριστώ πολύ, Σοφίλο Πρόεδρε. Birgit. Νομίζω ότι αν εξετάσουμε τα πρακτικά στοιχεία αλλά και το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να είτε ότι είναι εξαιρετική αυτή η απόφαση, είτε ότι είναι καταστροφική. Γιατί δεν ζούμε εν κενό, ζούμε μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν ας μιλήσουμε ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και μολονότι δεν ε, παραγνωρίζονται στην αξία και τη σημασία της διαφάνειας, δεν ξέρω πού ξεκινάει και πού τελειώνει αυτή θα τελειώσουμε με μια εντό αγωγικών διαφάνεια ε, και για τις ε, συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων ή των εθνικών αντιπροσωπιών. Δεν είναι σημαντικό κανείς να διαμορφώνει τη δική του θέση πρώτα πριν προχωρήσει σε συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τους άλλους. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Να μου πείτε ότι είναι απαραίτητο και σημαντικό για τον πολίτη να παρακολουθεί την νομοθετική διαδικασία. Είναι όντως νοητό ότι ο πολίτης μπορεί να καταλάβει και να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και τις αλλαγές στο κείμενο. Νομίζω ότι όποιος ενδιαφέρεται να καταλάβει τι εξέλιξη έχει ένα κείμενο, θα είναι ένας από τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους που ξέρουμε ότι ξεκίνησαν όλοι αυτοί, ξεκινούν μάλλον και μπαίνουν στη διαδικασία όχι την ώρα που έχει καταθέσει η Επιτροπή, τις προτάσεις της, αλλά την ώρα που τις σχεδιάζει στα σκαριφήματα ακόμα προσπαθούν να παρέμβουν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς και συμφέροντα. Και στις συζητήσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου μπορείτε να μου πείτε, αλλά δεν είναι ο κοινό πολίτης, είναι τα λόμπι, οι εμπλεκόμενοι φορείς και συμφέροντα. Επομένως εδώ δεν βλέπουμε τον ε, απλό πολίτη που ενδιαφέρεται για μια υπόθεση, αλλά κάποιον που θα έχει συμφέρον και που θα μπορεί ακόμα και όταν θα έχουμε πια ε, λάβει μια απόφαση στο Συμβουλίο του Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να παρέμβει και να επηρεάσει την κατάσταση. Ο απλός πολίτης συνήθως λέει, έχει βέβαια τη γνώμη του, αλλά λέει, εσύ ένα εξέλεξα, εσύ θα κάνεις τη δουλειά αν κοιτάξετε την κατάσταση πολλές φορές ε, σε ορισμένου φακέλους, είναι πολύ διαφορετική η εικόνα που βλέπουμε σε σχέση με το ενδιαφέρον των ομάδων πίεσης. Πολύ έντονη σε μερικές περιπτώσεις όπως μηδαμινή σε άλλες. Το είδαμε και με TTIP και με πολλά άλλα. Οι εμπλεκόμενοι, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα είναι αυτά που δείχνουν αυτό το ενδιαφέρον και όχι απλοί πολίτες. Και κάτι ακόμη που έχει πολύ μεγάλη σημασία την περίοδο που διανύουμε στην εποχή των ψευδών ειδήσεων η δουλειά του Κοινοβουλίου και κάθε Κοινοβουλίο κινδυνεύει να αλλάξει γιατί βεβαίως δεν είναι τίποτε το καινούριο οι ψευδείς ειδήσει, αλλά στην περίοδο, στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των μεσομασικής ενημέρωσης η διάδοση του είναι ραγδαία. Στη Γερμανία μπορώ να σας πω ότι είναι τόσο πολλά τα απροκάλυπτα ψέματα που διαδίδονται για να επηρεάσουν τον πολίτη που εγώ πια δεν είμαι σε θέση, δεν ξέρω τι να κάνω για να τα αποκρούσω όλα αυτά τα ψέματα. Η διαφάνεια λοιπόν, ναι, μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό, αλλά θα χρειάζεται να δίνουμε πάντα και το χρόνο για να αντιληφθούμε ποιος είναι αυτός που εκδηλώνει το ενδιαφέρον για την πληροφορία αυτή και πώς μπορούμε να το χειριστούμε το αίτημα. Τι σημαίνει το να του δώσουμε τη δυνατότητα της πρόσβασης. Τι συνέπειες θα έχει για τη δουλειά μας εδώ στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο. Και όπως είπα η απόφαση αυτή ούτε ιδανική είναι, ούτε καταστροφική. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση και βέβαια και σε σχέση με την επικοινωνιακή μας πολιτική. Ο πρόεδρος αγαπητής αν σιγά θα αρχίσουν να αποχωρούν οι συνάδελφοι Άρα καλό θα ήταν να βρούμε μια λύση, και αν θέλετε να απαντήσετε και εσείς στα σχόλια, με, τα, όλα όσα είπε η Μπιργκίτ και τα με τα επιχειρηματά σου, εγώ νομίζω ότι ως ΛΥΜΠΕ και ως Κοινοβούλιο θα πρέπει, το λέω έτσι αυθόρμητα, δεν μπορούμε εμείς, εμείς το Κοινοβούλιο ή η ΛΥΜΠΕ, να δώσουμε την εντύπωση ότι στρεφόμαστε κατά μιας απόφασης με μια έφεση, μιας απόφασης που ενισχύει τη διαφάνεια. Δεν θα φανεί καλό αυτό. Έτσι λοιπόν δεν θα πρότεινα να υποβάλουμε τέτοιο αίτημα στην ε, Επιτροπή Νομικής, Νομικών Υποθέσεων. Δηλαδή θα έλεγα να μην γίνει έφεση κατά της απόφασης, αν συμφωνείτε. Και αναλόγως να διατυπώσουμε και την ε, σύστασή μας προς τη Τζούρι. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό να δοθεί εντύπωση πως προσβάλλουμε την απόφαση με μια έφεση. Αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό και να δούμε και οι συντονιστές μετά τι θα πούνε για άλλες συστάσεις προς την Τζούρη. Ε, Θέλετε να πείτε κάτι ακόμα, έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Επιγραμματικά για τους κύριους Δε και Νετφέλτ και την κυρία Ζήπη. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Για να επανέλθω στα όσα είπατε. Χθε είχα την ίδια παρουσίαση στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων, όπου ορισμένοι βουλευτέ, είπαν πως έχει έντονα πολιτικό χαρακτήρο η απόφαση που θα λάβει η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων για την υποβολή έφεσης, για την άσκηση έφεσης. Δεν θα είναι μόνο δηλαδή νομική η απόφαση. Για το ζήτημα των ε, πιέσεων, των έξωθεν πιέσεων. Είναι σαφής η απόφαση όταν λέει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί πως ασκείται έξωθεν πίεση. Ανοίγει όμως τη δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα, προβλέπεται η δυνατότητα στον κανονισμό 1049, ότι δηλαδή αν υπάρχει πίεση που μπορεί να υπονομεύσει τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, και αυτό ακριβώς πρέπει να υπενήσετε το δικαστήριο. Λέει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορείς να επικαλεστείς το επιχείρημα της εξωθενπίεσης, αλλά θεωρητικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τώρα αν μου πείτε πώς θα πρέπει να διατυπωθεί ένα τέτοιο επιχείρημα, δεν ξέρω να σας το πω. Σε κάθε περίπτωση ίσως ξεχωριστά πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν έχω μια εύκολη και αυτόματη απάντηση. Θα πρέπει να το εξετάζουμε. Χρειάζεται περισσότερη μελέτη και επεξεργασία και κατεργασία η, η επιχειρηματολογία αυτή. Πολλά άλλα δεν έχω να πω για τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Αν όμως θεωρείτε ότι κάνω λάθος, πείτε μου. Ο πρόεδρος, όχι, οι ερωτήσεις όμως δεν ήταν ούτως ή ήταν ε, διαπιστώσεις από τους πεπειραμένους βουλευτές μας. Πάντως θα το προβλέψω, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε και για την ε, Γιούρη, ότι το βλέπει έτσι. Θα το προβλέψω στο, ε, στην ημερήσια διάταξη για τους συντονιστές. Και βεβαίως πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το θέμα την εικόνα που δίνουμε σε σχέση με τη διαφάνεια. Ξέρω, Μπιρκίτ, ότι δεν έχουν όλοι καταλήξει, αλλά εμείς στη ΛΥΜΠΕ πρέπει να δείξουμε μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της διαφάνειας. Δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι μας φοβίζει η αρχή της διαφάνειας ως αρχή. Πρέπει να είναι σαφές το, σαφές το μήνυμα που θα στείλουμε στην Γιούρη. Κυρία Ζήπλ, ε, εκτός μικροφώνου. Ναι, αλλά μπορεί να δοθεί αυτή η εντύπωση, συνεχίζει ο κύριος Μωρές. Πάντως καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Πρέπει να γίνει συζήτηση σε βάθος οπωσδήποτε. Και να κρατήσουμε και την επαφή με την Γιούρη σε όλη αυτή την υπόθεση, στην εξέλιξή της. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εκείνοι δεν έχουν ε, καταλήξει μια οριστική λύση. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο οποίο έχουμε σαφή, σαφέστατο και ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουμε. Για τα θέματα τα δικά μας. Ενώ η ΛΥΜΠΕ περισσότερο θα περιοριστεί στην, στα διαδικαστικά συστήματα. Την ουσία θα την κρίνουμε εμείς ως ΛΥΜΠΕ. Μπορεί να σας ε, ξανακαλέσουμε λοιπόν για το θέμα αυτό. Εγώ, όπως είπα, θα το περιλάω, θα το προβλέψω στην ημερησία της συνεδρίας των συντονιστών και σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.